Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία. Έχουμε έξι ψηφίσματα. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στον συνάδελφο Βανόρδεν για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, τα άτομα που ζουν στη Σρι Λάγκα έχουν uh, πληγεί και υποφέρουν τα τελευταία χρόνια λόγω των ε, τρομοκρατικών επιθέσεων. Σήμερα και η κυβέρνηση αλλά και ο λαός της Στριλάνκα χρειάζεται κατανόηση αλλά κυρίως υποστήριξη, βοήθεια από εμάς καθότι προσπαθούν να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους, να αποφύγουν την τρομοκρατία και να φτάσουν σε ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω ότι υπονοβεύοντας τις εμπορικές ε, συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τους βοηθάμε. Η καλύτερη στήριξη είναι οι εμπορικές συναλλαγές και όχι η so that there βοήθεια και υποστήριξη και νομίζω ότι το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να επαναφέρουμε αυτά τα άτομα, τους ε, Ταμίλ, και να τους βοηθήσουμε να μπορέσουν να επανενταχτούν και να ξαναζήσουν στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Βανόντεν. Ο κύριος Νταρόσα για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στηρίζω το ψήφισμα αυτό παρόλο που πιστεύω ότι δεν επικρίνει αρκετά αυστηρά την κυβέρνηση της Τριλάνκα. Όπως ξέρουμε, η πρόσφατη επίθεση τον τελευταίο καιρό κατά την άποψή μου με χιλιάδες νεκρούς ήταν ένα δείγμα ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Χιλιάδες πολίτες στη Σρι Λάγκα σήμερα ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες από υγειονομικής απόψεως με έλλειψη νερού και φοβερές δυσκολίες επιβίωσης. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να πιέσει από κάθε άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικά αλλά και πολιτικά, στην κυβέρνηση της Σρι εάν δεν υπάρχει απτή βελτίωση της κατάστασης. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την πίεση για να βελτιωθεί η κατάσταση των πολιτών της Λάκα και των Ταμίλ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ντερόσα. Ο κύριος Μάν για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά έχω, όχι ένα. Ο εμφύλιος πόλεμος που έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια φαίνεται να τελειώνει στη Σιλάνκα και από ό,τι καταλαβαίνω η κυβέρνηση η οποία σήμερα ελέγχει όλο το βόρειο τμήμα της χώρας, δεν έχει επιλύσει όλα τα προβλήματα, γιατί σήμερα τα πλήγματα δεν είναι μόνο πλήγματα του εμφύλου πολέμου, αλλά και φυσικές καταστροφές όπως το τσουνάμι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει κάποιες ε, από τις περιοχές, όχι μόνο την Σρι Λάνκα, αλλά και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Χρειάζεται όμως όχι μόνο οικονομική στήριξη, χρειάζεται μια στήριξη που να οδηγήσει στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα ξέρετε ότι υπάρχουν χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι, πρόβλημα όσον αφορά την υγειονομική υπερίσταληψη. τα φάρμακα, το πόσιμο νερό. Θα πρέπει λοιπόν, και αυτό είναι το προσυμφέρον και της κυβέρνησης να επιστρέψουν στα χωριά και στις περιοχές τους όλοι οι μετατοπιστέντες. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ εμείς μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να υπάρξει ελευθερία έκφρασης και ελευθερία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον τύπο. Δεν μπορεί πλέον να υπάρχουν φυλακισμένοι δημοσιογράφοι και δεν μπορεί η ελευθερία έκφρασης να έχει σαν αποτέλεσμα την κράτηση. Πιστεύω ότι η Σρι πρέπει να ξεκινήσει μια νέα κατάσταση. Πρέπει να δείξουμε επικοδομητικό πνεύμα, βεβαίως ε, καταπολεμώντας ε, την τρομοκρατία και τη βία. Χρειάζεται μια συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λιλάνκα έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα καθεστώς με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει επιτέλους αυτή η εμπόλεμη κατάσταση να πάει στο παρελθόν. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε κύριε Μαν, ο κύριος Χίγγινς έχει το λόγο. Η πολιτική απέναντι στους Ταμίλ από την κυβέρνηση της χώρας έχει καταλήξει σε μια φρίκη για, τους, για ε, της χώρας αυτές. Γίνονται επιθέσεις κατά ατόμων και ομάδων. Μετά από την ήττα λοιπόν των ε, τίγρων Ταμίλ ο εκφοβισμός συνεχίζει να υπάρχει στην χώρα αυτή. Υπάρχουν 205.000 άτομα τα οποία είναι κλεισμένα σε στρατόπεδα, ε, τα οποία εκφράζονται σε φορέ ανησυχίε για υπερβολικό συνοστισμό, έχουν ανεπαρκή πρόσβαση σε καθαρό νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και ιατρικές εγκαταστάσει που δεν υπάρχει, και εγκαταστάσεις που δεν υπάρχει ελευθερία. η κυβέρνηση του Ροτζιπάξη ε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια δικτατορία. Δράτω με τις ευκαιρίες που μας δίνετε σήμερα με το ψήφισμα για να καταδικάσω την κυβέρνηση. Έχω κάποιες φυλάξεις για την παράγραφο 4 που αναφέρει μάλλον ότι τα μύτη θα πρέπει να δισταθούν σοβαρά σε μια πολιτική ρύθμιση και να απαρνηθούν την τρομοκρατία και τη βία για πάντα. Πάντω η κυβέρνηση τη Σρι δεν είναι σε θέση να επιλύσει το πρόβλημα. Οι Ταμίλ έχουν δικαίωμα να αντιταχθούν σε, σε καταπίεση. Ο καλύτερο τρόπο για να του προσθέσουμε είναι ένα ε, αγώνα ε, κατά τη ε, κυβέρνηση του Σρι προκειμένου η κοινωνία της Σρι να μπορέσει να απελευθερωθεί από αυτήν την Χούντα. Χαίρομαι που μπορώ να συμφωνήσω με τις ε, επιτροπές οι οποίες καταδικάζουν το σοφινισμό της κυβέρνησης για τα δικαιώματα των Ταμίλ και για την αυτοδιάθεση του λαού Σρι Λάγκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Higgins κυρία Φανχάουτελα για 1,5 λεπτό. Όλα όσα είπαν οι συνάδελφοί μου σχετικά με την κατάσταση που κρατήσε στο Σρι είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε όταν η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρόσφατα οργάνωσε ακρόαση σχετικά με το όσα επικρατούν στην χώρα. Σχετικά με αυτόν τον εφιάλτη. Διαπιστώνουμε ότι οι 260.000 ε, άμαχοι Ταμίλ κρατούνται σε στρατόπεδο ε, παραβιάζοντας ε, κάθε δίκαιο. Η ελευθερία παρεμποδίζεται. Χθες μια οργάνωση που ονομάζεται ρεπόρτερ χωρίς σύνορα αναφέρουν ότι η Σρι Λάγκα βρίσκεται στην 62η θέση ανάμεσα σε 175 χώρες και στο ψήφισμα αυτό διαπιστώνουμε επίσης πως η οργάνωση των τοπικών εκλογών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε όλη φορά τώρα την εμπορική πολιτική, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το πώς η Σρι Λάγκα θα μπορέσει να υλοποιήσει τις απαιτήσει που περιέχονται στις διακηρύξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελπίζω η δουλειά να είναι αντικειμενική προκειμένου από τα συμπεράσματα να γνωρίζουμε κατά πόσον η Σρι Λάγκα αξίζει αυτού του γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων. Ευχαριστώ κύριε Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Χάουταλα. Καταρχήν το κύριο Σπόσελεξ, ο νόμο των πολιτικών ομάδων. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πραγματικά ότι στη Σρι Λαγκά πολλά γεγονότα δεν είναι ακόμα γνωστά. Όπως ξέρετε, πρόκειται για μία κλιμάκωση ενός προβλήματος που αρχικά ήταν πρόβλημα εθνοτήτων. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι των οποίων τα νόμιμα δικαιώματα δεν έχουν πλέον αναγνωριστεί ακόμα και εγγυηθεί. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια πολιτική λύση. Όντως, σήμερα η βία έχει καταπολεμηθεί. Όμως, οι αιτίε αυτών των συγκρούσεων αυτής της διαμάχης, δυστυχώς, δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Είναι πιο εύκολο να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά όπως ακριβώς έγινε και στη Βοσνία, ο πόλεμος σταμάτησε, λύση δεν έχει βρεθεί. Για να υπάρξει λοιπόν σταθερότητα θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα των μειονοτήτων που υπάρχουν εδώ και αιώνες. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να παίξουμε ένα μεσολαβητικό ρόλο έτσι ώστε να σταματήσει η πραγματική αιτία των προβλημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκίλτα Φον Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται ένα χρόνο μετά την ήττα των ε, τίγρεων τα μήλα, ότι δεν έχουν σταματήσει τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Για το λόγο αυτό ξέρουμε ότι οι αρχές ε, κρατούν σε στρατόπεδα περισσότερο από 250.000 άμαχους τα μήλ. Ξέρουμε ότι και κάποιος η κράτηση και κάποιου δημοσιογράφου και η επιβολή ποινή πάνω από 20 χρόνια για συμμετοχή διαδηλώσεις είναι κάτι το οποίο καταδικάσαμε. Εάν ήταν ε, μέλος, αν είχε προσυπογράψει μάλλον στη σύμβαση της ε, ΟΤΑΒΑ η χώρα αυτή, δεν θα υπήρχαν προβλήματα. Οι κάτοικοι της Σρι Λάγκα πραγματικά αξίζουν καλύτερη ζωή και δημοκρατία. Ευχαριστώ, πολύ τη συνάδελφο, η κυρία Ντέλη. Monsieur Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, εδώ και μήνες η κυβέρνηση Σρι δεν λέει τίποτα όσον αφορά το θέμα των Ταμίλ και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν φυλακισμένοι εδώ και δύο χρόνια και παραβιάζονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των φυλακισμένων. Όπως ξέρετε, πάνω από 280.000 φυλακισμένοι κρατούντο στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού από την κυβέρνηση. Μπορούσαν να εγκαταλείψουν τα στρατόπεδα κράτησης ακολουθούμενοι από στρατιωτικούς μόνο σε περίπτωση που έπρεπε να νοσηλευθούν σοβαρές επιδημίες, δυσεντερία και άλλες πλήττουν τα άτομα αυτά. Πάνω από 100.000 ε, πρόσφυγες στα ΜΟΥΛ επρόκειτο να ελευθερωθούν και η πίεση θα πρέπει να συνεχιστεί προς την κυβέρνηση Ιρλάνκα ώστε να απελευθερωθούν όλοι οι φυλακισμένοι, να αφαιθεί ελεύθερη πρόσβαση στους δημοσιογράφους και να σταλεί ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ντέλη και τώρα η διαδικασία Catch the Eye. Εκπρόσωπος του Λονδίνου που ήταν πάρα πολλές φορές πόλη που υπέστη τρομοκρατικές ε, ε, δραστηριότητε, ε, είμαι αλληλέγγυος προς τα δικαιώματα των Ο πρόεδρος Ρότζερ Παξ είναι δημοκρατικά εκλεγμένος και θα θέλαμε να τον ε, βοηθήσουμε για να μπορέσει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν ε, δικαστούν οι υπεύθυνοι των τρομοκρατικών εκδηλώσεων από τα δικαστήρια, νομίζω ότι θα έχουμε να κάνουμε με μία επιτυχία της κυβέρνησης Είμαι πεπισμένος ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να εγγυηθούμε ότι η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της ε, Σρι πρέπει να προστατευτεί για να έχουμε σύντομα μια χώρα η οποία θα μπορέσει να αναπτυχθεί σύντομα. Και βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουν οι αθώοι να γυρίσουν στα σπίτια τους. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως Ιρλανδός εκφράζω την ικανοποίησή μου για το ότι οι συνάδελφοί μου ανέφεραν όλους τις ανησυχίες τους σχετικά με τη Σρι Λάγκα. Η Ιρλανδία θα πρέπει να ασχοληθεί με το ζήτημα διότι βλέπουμε ότι και στο παρελθόν στην Ιρλανδία υπήρχαν διακρίσεις και χανόντουσαν ζωές και τελικά καταλήξαμε σε συζητήσεις, διαπραγματεύσεις κλπ. Και, και επιλύθηκε το πρόβλημα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει ένα νέο καθεστώς στο οποίο ο Πρόεδρος ε, θα πρέπει να συμμετάσχει και να φροντίσει να προωθήσει την ε, ειρήνευση, τη συμφιλίωση. Όλα αυτά φυσικά θα πρέπει να ε, έχουν ως αποτέλεσμα την επιστροφή στην δημοκρατική διαβίωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κορόλα. Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθήσαμε τι εξελίξει στη Σρι Λάγκα επανειλημμένα και κάθε φορά χάναμε κάθε ελπίδα για την εξέβριση λύσης. Ο πόλεμος διήρκησε 25 χρόνια, αλλά επιτέλους ε, έλαβε τέλος μετά από τις πρόσφατες εξελίξει. Αυτό όμως οδήγησε σε πάρα πολλή δημιουργία πολλών προσφύγων ε, και καταπάτηση δημοκρατικών δικαιωμάτων. Στα στρατόπεδα υπάρχουν άτομα τα οποία υποφέρουν, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα. Ελπίζουμε πως οι αρχές ε, θα μπορέσουν να λάβουν και να προωθήσουν την ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε ανάγκη επίση ε, να αναλάβει τις ευθύνες της η διεθνής κοινότητα για να οικοδομήσουν ξανά ένα δημοκρατικό αθεστώς. Επίση πρέπει να δοθεί βοήθεια για την εξουδετερήση των αρκοπαιδίων. Ο κύριο Ρόμβα είχε έχει το λόγο. Θα ήθελα να λάβω το λόγο πρώτα απ' όλα για να τονίσω αυτό που είπε η συνάδελφο Χάουταλα, ότι δηλαδή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο ΙΕ σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο ο Ερθρό Σταυρό, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη. Θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτό που είπε ο συνάδελφο Βανόβδο, διότι θεωρώ ότι δεν είναι ορθό εάν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σαφές μέσο όπως η, ε, το σύστημα γενικημένων προτιμήσεων για να ε, ε, εκμεταλλευτούμε την κατάσταση. Όχι, δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε εάν οι αρχέ τη ΛΑΝΚΑ αυτή τη στιγμή πράττουν τα απαραίτητα προκειμένου να ενσωματώσουν τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην νομοθεσία του. Αυτό είναι απαραίτητο να απαιτηθεί από την ε, διεθνή κοινότητα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μην ανανεωθούν οι γενικευμένε προτιμησιακέ συμφωνίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Όρμπαν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, το ζήτημα μας από σχολή είναι η κατάσταση στη Σρι Λάγκα. Ξεκινήσαμε με την κυβέρνηση τη Σρι Λάγκα έναν διάλογο προκειμένου να θέσουμε τις βάσεις για μια νέα σχέση όπου και οι δύο πλευρές θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για να καταλήξουμε στην επίλυση των προβλημάτων που μας απασχολούν σήμερα. Μας ενισχύει ιδιαίτερα η ανθρωπιστική κατάσταση η οποία είναι κρίσιμη στα στρατόπεδα όπου οι πολίτες οι οποίοι έχουν ε, εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας ε, κρατούνται. Η παραμονή αυτών των ανθρώπων στα στρατόπεδα αποτελούν παραβίαση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα κατάφορη. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε όλα αυτά τα άτομα να ε, έχουν ελεύθερη διακίνηση αλλά και την άμεση πρόσβαση στα στρατόπεδα των ε, υπευθύνων των ανθρωπιστικών, της ανθρωπιστικής βοήθειας και η Κομισιόν επίσης ε, ανησυχεί για τα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Σρι Λάγκα. Έχουμε λάβει πολλές προφορίες ε, αναφορικά με κάποιες καταδίκες, απαγωγές ε, και εκφοβισμούς αλλά και εκβιασμούς. Ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα σε ό,τι φορά τη συμφιλίωση στην ίσο και αυτό θα συνεχιστεί εάν δεν ληφθούν απόψη η κατάσταση των Ταμίλ και όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η διαδικασία συμφιλίωσης θα πρέπει να περάσει μέσα από την συνεργασία των κομμάτων. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια μελέτη για την κατάσταση των δικαιωμάτων στην Στριλάνκα. Λάγκα. Στόχος αυτής της μελέτης που βασίστηκε σε μια αποστολή είναι του κατά πόσον η χώρα πληρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει όταν της παρασχέθη η βοήθεια για την καλή διακυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση το σύστημα γενικημένων προτιμήσεων Plus μετά από αυτήν την έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε πάρα πολλές ελλείψεις ε, και μάλιστα πολύ σοβαρές σε ό,τι αφορά τρεις ε, συμβάσεις ε, των Ηνωμένων για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη Διεθνή Σύμβαση για τα πολιτικά δικαιώματα και τα αστικά δικαιώματα, τη Σύμβαση κατά των βασανιστήριων και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Κάτι το οποίο δείχνει πως τη στιγμή αυτή η Σρι Λάνκα δεν εφαρμόζει αυτές τις διεθνείς συμβάσεις και είναι αναπόφευκτο η κατάσταση αυτή να επηρεάσει τις ε, εμπορικές ε, σχέσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας ε, SPG+. Διότι όλοι οι δικαιούχοι αυτής της συμφωνίας θα πρέπει να έχουν κυρώσει και να εφαρμόσει όλες αυτές τις συμφωνίες τις οποίες προανέφερα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο Όρμπαν. Τέλος της συζήτησης και θα ψηφίσουμε αμέσως. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι στις επεξηγήσεις ψήφου και κατά την διαδικασία Catch the Eye εξαντλήσαμε την διαδικασία αυτή. Πλέον δεν